ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα, την πρόσφατη ανακοίνωση, θα δείτε ότι μιλεί πολύ για ανταγωνιστικότητα, για προστασία των Ευρωπαίων γεωργών, για κλιματικές αλλαγές, αλλά δεν αναφέρεται σχεδόν καθόλου σε θέματα ανάπτυξης. Αυτά για τις γεωργικές επιδοτήσεις. Οι συστάσεις μας προκύπτουν λοιπόν από αυτά που είπα, ενίσχυση στην συζήτηση περί κοινής αγροτικής πολιτικής των πτυχών ανάπτυξης, κατάργηση των επιστροφών εξαγωγών. Αυτό ίσως γίνει ούτως ή άλλως όταν θα ολοκληρωθεί ο γύρος της Ντόχα. Αλλά επί του παρόντος δεν διαφαίνεται πότε θα γίνει αυτό. Και επίσης όταν θα γίνει η αναθεώρηση της ΚΑΠ θα πρέπει να εξεταστούν ποιες είναι οι επιπτώσεις και στο μέλλον των διαφόρων επιδοτήσεων. Κάτι διαφορετικό τώρα, αλλαγή κλίματος πάλι είδαμε εδώ και ε, φωτεινά σημεία και λιγότερο φωτεινά. Για τα φωτεινά σημεία είναι η ανάπτυξη της, ε, μάλλον η εξέλιξη της ε, πολιτικής για την προστασία του κλίματος, ή από τις αλλαγές του κλίματος, έχει λάβει κυρίαρχη θέση στην, στις τρέχουσες συζητήσεις και στη συνεργασία και στις χρηματοδοτήσεις όπου ε, τα κονδύλια που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η DREF που είναι το Παγκόσμιο Ταμείο για την Συνεργασία για την Ανάπτυξη. Γίνεται λοιπόν αυτή η συνεργασία, γίνονται και προσπάθειες από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειωθούν οι εκπομπές ε, αερίων του θερμοκηπίου και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό και οι επιπτώσεις στην, στις αναπτυσσόμενες χώρες και για τις εκτός μάλλον σε τις χώρες. Εν τέλει, κάποια πρόοδος έχει γίνει και σε σχέση με τα έγγραφα για τις θετικές των χωρών και την συμπερίληψη των πτυχών της αλλαγής του κλίματος σε αυτά. Έχω εξετάσει καμιά δεκαετία από τα έγγραφα αυτά και βλέπω ότι η κλιματική αλλαγή αναφέρεται σε πολλά από τα έγγραφα αυτά, αν και όχι σε όλα. Έρχομαι τώρα στις λιγότερο φωτεινές πτυχές, ας πούμε έτσι. Κάποια πρόοδο έχει γίνει ή γίνεται για την ένταξη της κλιματικής αλλαγής στον σχεδιασμό της ανάπτυξης, ακόμα όμως δεν έχει επιτευχθεί παντού, δεν έχει περιληφθεί δηλαδή παντού. Είπα τέλος ότι αυξανόμενη χρηματοδότηση διατίθεται για θέματα μετριασμού και προσαρμογής, ε, στις αλλαγές του κλίματος δηλαδή, αλλά σε σύγκριση με τα απαιτούμενα ποσά παγκοσμίω, αλλά και ποιο θα ήταν, ε, ε, ποια θα ήταν δίκαιη κατανομή ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει φτάσει στα επίπεδα αυτά. Δεν είναι μόνο το πρόβλημα με τη χρηματοδότηση, ότι δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση, ότι δεν είναι αρκετά προβλέψιμη, ότι δεν παρακολουθείται επαρκώς. Υπάρχουν και ορισμένα έργα, για παράδειγμα ε, μεγάλες εγκαταστάσεις καύση στην Νότια Αφρική που υποτίθεται ότι έχουν διπλή χρήση, δηλαδή και παραγωγής ενέργειας, ε, είναι αμφισβητούμενα και όταν συνομιλεί κανείς με ανθρώπους των Υπουργείων, για παράδειγμα στην Ομοσπονδιακή Γερμανία, βλέπω ότι μένουν πολλά ανοιχτά ερωτήματα, δηλαδή πώς θα πρέπει να γίνει η προσαρμογή στι αναπτυσσόμενες χώρες, γιατί πολύ συχνά Υπάρχουν έργα αναπτυξιακά που θα βοηθήσουν ε, τους ανθρώπους να βγουν από τη φτώχεια και να μεταφέρουν και κάποια τεχνογνωσία. Αυτά είναι και καλά προγράμματα για την προσαρμογή. Είναι λοιπόν το θέμα να αναζητηθούν τα σωστά έργα. Οι συστάσεις τώρα για την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να είναι να αναχθεί η κλιματική αλλαγή έστω να περιληφθεί σε όλα τα έγγραφα να υπάρξουν κατευθυντήρες γραμμές για την ευρωπαϊκή βοήθεια που πρέπει να είναι λεπτομερής. να γίνεται climate screening για, όλες τις, ε, για όλα τα μελλοντικά έργα. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να εφαρμοστεί. Σε σχέση με τη χρηματοδότηση, η χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι προβλέψιμη, μακράς διάρκειας, επαρκής και βεβαίως να παρακολουθείτε, να υπάρχει monitoring δηλαδή. Γιατί για την ώρα υπάρχει σύγχυση ποια χρηματοδότηση έχει σχέση με την προστασία του κλίματος και ούτε καθεξής. Είναι δηλαδή ε, τα πράγματα εκεί κάπως ασαφή. Και εν τέλει να διασφαλιστεί ότι χρηματοδότηση ευρωπαϊκή δεν δίνεται για έργα DHD σε αναπτυσσόμενες χώρες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχουν τώρα τα μέλη της Επιτροπής μας. Θέλει κάποιος, ο κύριος Μίτσελ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ο κύριος Μίτσελ Γαλλικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα, τις τόσο ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα ε, να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος της συναδέλφου που ε, δεν θα μπορέσει να έρθει σήμερα εδώ και θα μιλήσω εγώ στη θέση της ε, όσον αφορά το θέμα της διατροφικής ασφάλειας. Διάβασα τον κανονισμό και εκπλήσωμαι που η Ταϊλάνδη η οποία ε, ε, ε, είναι η μεγαλύτερη παραγωγός ας πούμε ε, τροφίμων και τροφών στην περιοχή. Έχει γειτονικέ χώρες όπως η Βυρμανία που πραγματικά μαστίζεται από λοιμό. Τι μπορεί να γίνει σε τοπικό επίπεδο έτσι ώστε χώρες όπως η Ταϊλάνδη ας πούμε να είναι εταίρος μας αλλά ταυτοχρόνως να βοηθάει και την ε, περιοχή. Έχουμε ε, οικοδομήσει τέτοιου είδους εταιρικέ σχέσεις. Δεύτερον, σε σχέση με το εμπόριο. Μελετήσατε το ενδεχόμενο ε, και την δυνατότητα άειλων αγαθών που θα εμπορεύονται ή χρηματοπιστωτικών ας πούμε συναλλαγών. Μίλησα πρόσφατα με την Υπουργό Οικονομικών της ε, Ρουάντα που είναι ε, από τους ε, εταίρους μας στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Και Ε, μου έλεγε την δυνατότητα οι κάτοικοι και οι γεωργοί να μπορούν να υποθηκεύσουν κατά κάποιο τρόπο αυτή τη βοήθεια έτσι ώστε να έχουν ένα αντικείμενο εμπορίας. Στη σελίδα 27 αναφέρεται ότι οι γεωργικές επιπτώσεις έχουν ε, κυρίως αρνητικό ε, έχουν αρνητική επίπτωση στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ενώ σελίδα 21 λέτε ότι ε, θα πρέπει να μελετηθεί το σύστημα των γεωργικών επιδοτήσεων έτσι ώστε να δούμε εάν υπάρχουν κερδισμένοι ή χαμένοι και ποιοι είναι αυτοί. φαίνεται ότι υπάρχουν έτσι κάποιες αμφιλεγόμενες αποχρώσεις. Και τελευταία ερώτηση, μιλώντας για εμπόριο. Έχετε μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο ε, ο αναπτυσσόμενος χώρο, οι αναπτυσσόμενες χώρες μπορούν ή θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ε, μια αγορά όσον αφορά το εμπόριο ε, διοξιδίου του άνθρακος. Τρεις ερωτήσεις και μετά θα απαντήσετε. Η κυρία Κέλλερ. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις που τις βρήκα πολύ ενδιαφέρουσες. θέσατε τον δάχτυλο σε πολλά προβλήματα που θεωρούμε ότι είναι κρίσιμη σημασία αν θέλουμε να επιτύχουμε την ανάπτυξη. Πάντοτε λέμε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει συνοχή και όχι να παίρνουμε με το ένα χέρι αυτά που δίνουμε με το άλλο. Η έκθεσή σας λοιπόν, η παρουσία σας δείχνουν ότι έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε για να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο. Τώρα που έχουμε τη μελέτη αυτή, νομίζω πρέπει να σκεφτούμε ως Επιτροπή Ανάπτυξης με ποιον τρόπο θα εφαρμόσουμε τα συμπεράσματα αυτά, πώς θα τα περιλάβουμε στις επόμενες εκθέσεις μας που θα γράψουν οι συνάδελφοί μας. Και για τις γνωμοδοτήσεις που πρόκειται να συντάξουμε για το γενικευμένο σύστημα προτιμήσεων. Αυτό που βρίσκω λυπηρό είναι ότι στο θέμα αυτό δεν είμαστε εμείς η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, διότι ναι μεν είναι θέμα ε, χρηματοδοτικό, αλλά είναι και θέμα κυρίως πρωτίστως ανάπτυξης. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα όσα είπατε βεβαίως. Λέτε ότι η αναθεώρηση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να κάνουμε μια καλύτερη σε βάθος μελέτη του τι σημαίνει αυτή η διάβρωση των προτιμήσεων. Διότι προβάλλεται το επιχείρημα πάντοτε ότι θα υπάρχει λιγότερη, λιγότερος ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών GSP αλλά και των ΕΠΑ. Διάβασα ωστόσο ένα άνθρωπο που λέει ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των ομάδων αυτών χωρών αφού το εμπόριό του αφορά άλλα προϊόντα. Αν λοιπόν δεν υπάρχει ανταγωνισμός, τότε δεν υπάρχει και ε, ε, όφελος για τις χώρες ΕΒΑ. Για την μετανάστευση, συμφωνώ μαζί σας ότι είναι δύσκολο, ακαθόδες θέμα. Πώς εντάσσεται στην οχή δεν είναι σαφές για μένα, διότι φαίνεται να υπάρχει επιθυμία να συνεχιστούν να δίνονται χρήματα από τα Ταμεία της Ανάπτυξης για να κρατηθούν οι μετανάστες στις πατρίδες τους. αλλά και στην διαδικασία αναθεώρησης του προγράμματος, του θεματικού προγράμματος μετανάστευσης, ίσως υπάρχει η δυνατότητα να ασκήσουμε κάποια επιρροή, αφού είναι από τα πιο σημαντικά ζητήματα, όπου βλέπουμε να υπάρχουν ασυνέπειες, αλλά δεν υπάρχει νομίζω πολιτική βούληση για να αλλάξουν πολλά πράγματα. Για τη γεωργία, η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Κομισιόν κάνει τώρα μια μελέτη αντικτύπου για πέντε περιπτώσεις από την Αφρική και αυτό είναι καλό διότι ακούσαμε πριν από την Επίτροπο ότι η κοινή αγροτική πολιτική δεν έχει καμία σχέση με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Φαίνεται ωστόσο ότι αλλάζει κάπως η νοοτροπία αυτή και στην Επιτροπή. Πάντως πρέπει να παρακολουθούμε προσεκτικά την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η αναθεώρηση της ΚΑΠ. Για την κλιματική αλλαγή νομίζω δεν αναφερθήκατε στα βιολογικά καύσιμα, τα οποία αναφέρει η Κομισιόν ως θετικό ε, παράδειγμα ανάπτυξης στα έγγραφά της, όπως είπα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διερωτώ αν βλέπετε κι εσείς κάποια φωτεινά σημεία ε, στην πολιτική συνοχή για το θέμα αυτό. Και τελευταία παρατήρηση είπατε στην μελέτη σας ότι η υπόθεση της παρούσας επιτροπής ότι φθηνά αγροτικά προϊόντα κατακλείουν τις αναπτυσσόμενες χώρες διότι λέτε ότι οι χώρες αυτές έχουν υψηλούς δασμούς, φαίνεται πως αυτή η υπόθεση θεωρείται ότι είναι εσφαλμένη. Εμείς παράγουμε υπερβάλλον εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καταλήγει στην Αφρική, για παράδειγμα. με ένα αγρόκτημα που εκτρέφει κοτόπουλα. Και το βασικό μέρος του σώματος του πουλιού μένει στην Ευρώπη για κατανάλωση και τα λιγότερο ε, σημαντικά και φθηνά καταλήγουν στην Αφρική για κατανάλωση. Δεν νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να εξετάζουμε μοναχά τους δασμούς υπάρχουν και άλλες πτυχές του ίδιου θέματος ε, της εξαγωγής δηλαδή γεωργικών προϊόντων. Σας ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup. Ευχαριστώ. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Γκριμούν. Avec votre permission. Εάν ε, μου επιτρέπετε κυρία Πρόεδρε, θα... είμαι συνεργάτης του κυρίου Γκριμό και θα απαντήσω εγώ. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για αυτή την συζήτηση και αυτές τις παρουσιάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και κέρδιες γιατί έρχονται σε ε, μια στιγμή που ακριβώς δουλεύουμε πάνω στην συνοχή των πολιτικών ανάπτυξης. Αυτά που αναφέρετε είναι πολύ ενδιαφέροντα κατά την απόψή μας διότι συχνά ε, διαπιστώσαμε ότι είναι σημεία τα οποία και εμείς έχουμε ε, θίξει στις εκθέσεις Επιτροπής όσον αφορά ε, τις ελλείψεις των πολιτικών από το 2010 μέχρι το 2013. Ενδεχομένω ε, θα πρέπει να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε μερικά θέματα. Βεβαίω, ε, τα εμπορικά ε, ζητήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Οι χώρες που εντάσσονται στο σύστημα, στο γενικευμένο σύστημα προτιμήσεων μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ και θα τι μελετήσουμε εντελεχώς. Όσον αφορά την γεωργική πολιτική. Είναι γεγονός ότι η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας έχουν ζητήσει έκθεση ε, για να μελετήσουν τις επιπτώσεις μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Ε, ολοκληρώνεται όπου να είναι η μελέτη αυτή και με τον τρόπο αυτό θα ολοκληρωθεί και η μελέτη επιπτώσεων ε, της μεταρρύθμισης στην γενικότερη αναπτυξιακή ε, πολιτική. Θα δείτε τα αποτελέσματα όταν δημοσιευθούν. Όταν ε, ε, σε σχέση τώρα με την πολιτική μετανάστευσης βεβαίως δουλεύουμε στενά με την Γενική Διεύθυνση HOME. Νομίζω ότι έχει υπάρξει κάποια τροποποίηση όσον αφορά τη στάση των υπαλλήλων σε σχέση με τα όσα αναφέρονται στην έκθεση, γιατί ε, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή εμείς επικεντρώνουμε την προσπάθειά μας στον ίδιο το μετανάστη. Αναπτύσσουμε ε, συστάσεις πολύ συνεκτικές με άλλες πολιτικές, έτσι ώστε να έρθουμε σε επαφή και με την διασπορά των χωρών και να μην εστιάσουμε μονάχα την ελεγχιστοποίηση ε, των μεταναστευτικών ρευμάτων σε σχέση με τις ίδιες τις χώρες από τις οποίες αυτά ε, προέρχονται. Επίσης ε, υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο που έχει σταλεί στις χώρες μέλη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της έκθεσης του 2011 και ελπίζουμε ότι θα μπορούμε να έχουμε πολύ πιο συγκεκριμένε απαντήσει την επόμενη φορά που θα συναντήσουμε το Κοινοβούλιο όσον αφορά αυτή την έκθεση του 2011. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στι ε, εμπειρογνώμονέ μα. Θα ξεκινήσω με την πρώτη ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ για τι ερωτήσει σα. Θα αρχίσω από το τέλος. Χαίρομαι πάρα πολύ για την ερώτηση εκείνη που αφορούσε για το τι γίνεται με τις αγροτικές επιδοτήσεις αντισόμενες χώρες και ποιες είναι οι συνέπειες όσον αφορά τις χώρες που εξετάζουμε. Και αυτό θέλησα να τονίσω στην έκθεση ότι κατά κοινή ομολογία στρεβλώνονται το εμπόριο από τις επιδοτήσεις. Και θεωρούμε ότι η κατάργηση των επιδοτήσεων θα ωφελήσει και τους μεν και τους δε, αναπτυσσόμενους και ανεπτυγμένους. Δεν μπορώ να το εξηγήσω λόγω πίεσης χρόνου στην εισήγηση. Να δούμε τώρα κατά πόσον έχουμε αντίφαση. Δεν έχουμε αντίφαση στο κείμενο, διότι οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν πολλές διαφορές μεταξύ τους. Και αυτό που θέλω να σας τονίσω είναι το ότι αυτές οι χώρες ωφελούνται από τις ε, ενισχύσεις αυτές. Υπάρχει ένα θέμα διαφοράς της παγκόσμιας τιμής και τιμής της Ευρωπαϊκής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε, τελικά, μπορούν να εισαγάγουν φθηνότερα οι χώρε αυτέ. Άρα ωφελούνται και ω εξαγωγή και ω εισαγωγή και έτσι ωφελούνται οι καταναλωτέ. Επίση είναι σημαντικό το να το μελετήσουμε και ω επομένω καταναλωτέ και όχι μόνο ω εξαγωγή. Έτσι να δούμε το τι γίνεται με τι χώρε αυτέ. Βέβαια θα πρέπει να υπάρχει μια περίοδο προσαρμογής για αυτούς που ζημιώνονται. Αυτοί πάντως που τώρα θεωρούνται ότι ζημιώνονται, αύριο θα είναι εντάξει, γιατί έχουν το πλεονέκτημα για τις εξαγωγές, όπως οι χώρες της ομάδας Κάρνς. Βραζίλια, η ΙΠΑ, χωρίς βέβαια η να είναι ανοσόμενη χώρα, όμως θα ωφεληθούν και εκείνοι. Αλλά και οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα ωφεληθούν από την κατάργηση των ενισχύσεων επομένως, συνολικά να δούμε το ότι θα πρόκειται για διορθωτική κίνηση εάν γίνει αυτή η κατάργηση. Όσον αφορά τώρα τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ΑΣΕΑΝ δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη μελέτη για αυτόν τον τομέα και για συγκεκριμένε χώρες. Όμως πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο θέλει να προβεί σε περαιτέρω απορριθμίσει η Ένωση. Έχουμε κάποιες συμφωνίε ελευθέρω εμπορίου, καλύπτουν και τέτοιες υπηρεσίες. Άρα με τις διάφορες συμφωνίες ευθερόμπαριου θα καλυφθεί ο τομέας των υπηρεσιών αυτών, των χρηματοπιστωτικών. Τώρα, θα ήθελα να σταθώ στο θέμα των προτιμήσεων. Πάλι δεν σας τα είπα αναλυτικά λόγω ποιης χρόνου στην εισήγηση, γιατί από το σύστημα γενικευμένων προτιμήσουν, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται, πώς εξελίσσεται, πώς εξελίσσονται οι δασμοί, τι γίνεται με, τις, ε, με τους διαφορούς γύρους και διαπραγματεύσεων. Άρα υπάρχουν μελέτες που λένε ότι όταν ε, έχουμε μικρό περιθώριο προτίμησης, τότε εισαγωγές εξαγωγές δεν ωφελούνται, δεν ασχολούνται, δεν έχει ενδιαφέρον το να ασχοληθούν με την ε, προτίμηση. Δεν άξιζε τον κόπο επομένω. Τι εγκαταλείπουν τις προτιμήσεις. With regards to other questions. Άλλες ερωτήσεις είχαμε θέμα. Καλά. Να συνεχίσουμε τώρα με τις άλλες ερωτήσεις που επευλήθησαν. Ο κύριος Μίτσελ έχει υποβάλει κάποιες ερωτήσεις. Κάτι λέγατε για ιδιοκτησία. Όσον αφορά την εμπράγματη ιδιοκτησία, μας είπατε χτες. Και επίσης αυτή την ενημέρωση για αυτά τα δικαιώματα. Αυτά τα δικαιώματα είναι δυνατόν να αποτελέσουν τμήμα τη στρατηγική κατά τη φτώχεια. Θα πρέπει να συμπληρωθούν και από άλλε πολιτικέ. Αυτά συζητούσαμε. Δεν είναι πανάκια τα μέτρα, τα δικαιώματα αυτά. Άρα, επομένως, υπάρχουν και εναλλακτικές. στην αγορά των εκπομπών διοξιδίου. Η Παγκοσμία Τράπεζα ασχολείται, στηρίζει τις αντισόμενες χώρες. Τώρα κατά πόσον αυτό μακροπρόθεσμα θα ωφελήσει την ανάπτυξη, αυτό ακόμα δεν έχει κρυφθεί οριστικά. Αναφέρθηκε χθε κάτι σχετικά το οποίο μας οδηγεί στην προβληματική για τα βιοκάψιμα, Αυξάνεται η ζήτηση. Όσον αφορά δηλαδή την ε, ε, απόκτηση ακινήτων ε, γης σε μεγάλη κλίμακα στις αντισόμενες χώρες. Βλέπουμε ότι και εδώ τα πράγματα δεν έχουν αποκρισταλωθεί. Ε, υπάρχουν διάφορα μέσα πολιτικής για την καθαρή ανάπτυξη για τα προϊόντα CDM. Άρα, θα πρέπει οι επενδύσεις να γίνονται με τον πιο σωστό τρόπο, ούτως ώστε να ωφεληθούν οι χώρες. Προς το παρόν όμως το τοπίο δεν είναι και τόσο αισιόδοξο. Οπότε και εμείς με αυτό ασχολούμαστε σε αυτό το ενημερωτικό σημείωμα. Άλλες ερωτήσεις. Βλέπω ότι το μέλλον της ΚΑΠ εξετάζεται σε σχέση με την αναπτυξιακή πολιτική. Αυτό είναι πολύ θετικό σίγουρα. Επίσης, τα βιοκαύσιμα εδώ υπάρχει συνέπεια στις πολιτικές μας, παρά το το θέμα είναι τόσο διφορούμενο. Και έχω μελέτες για το ότι η ενασχόληση και παραγωγή βιοκαυσίμων έχει οδηγήσει στο να χάσουν σε εκμεταλλεύσει τους πολύ γεωργοί, το οποίο δεν είναι θετικό. Άρα να γίνεται κάτι σε τοπική κλίμακα, να εμπλέκονται οι τοπικοί και άρα να βγαίνει κάτι θετικό για αυτούς τους φουκαράδες που είναι φτωχοί άνθρωποι όμως πολλά εξαρτώνται κάθε φορά από τις ε, ε, περιστάσεις, τις συνθήκες Οπότε ακριβώς το θέμα είναι αυτό, ο ανταγωνισμός ε, παραγωγής και βιοκαυσίμων. Το συζητήσαμε χθε. Οι υψηλοί δασμοί. Και η αγορά ειδών διατροφής στις αμπλησόμενες χώρες. Οι εθνικέ κυβερνήσει των χρόνων αυτών πρέπει να λάβουν κάποια μέτρα και και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι μπορεί να κάνει. Ούτω ώστε να τι θα σέψουν τι εξελίξει και μην τα κάνει όλα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια δεν εξαρτώνται τα πάντα από τους δασμού, Αλλά θα πρέπει όλε οι πλευρέ να προσπαθήσουν. Αυτά. Ελπίζω ότι απάντησα όλα όσα με αφορούσαν από τα ερωτηθέντα. Ελπίζω ότι σας κάλυψε Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η κυρία Κέλλερ όμως έχει ερώτηση. Σε σχέση με αυτά που είπατε, Βεβαίω και θα πρέπει οι κυβερνήσει των να κάτι να κάνουν. Αλλά και εμείς θα πρέπει κάτι να κάνουμε Τώρα, όσον αφορά την περικοπή των ε, γεωργικών ενισχύσεων, είπαμε ότι σε πρώτη φάση, αν κατάλαβα καλά, θα φύγουν οι καταναλωτέ τη χώρε. Στην πρώτη φάση. Επίση, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με εκείνου που καταναλώνουν και δεν προβληματίζονται σε σχέση με το εισόδημα και την πηγή του. Όμως αυτοί που παράγουν τα γεωργικά προϊόντα και τα που πολλούν, ε, θα πρέπει να μπορούν να παράγουν περισσότερα, καλύτερες τιμές και να μην ε, πέφτουν έξω και να χάνουν την εκμετάλλευσή τους. Επομένως, βλέπουμε πώς επηρεάζεται το εισόδημα αυτών των ανθρώπων και πώς καταπολεμείται η φτώχεια. Να δούμε δηλαδή τον όλο κύκλο, το ότι ο καταναλωτής δεν είναι ο καταναλωτής, είναι και παραγωγός ταυτόχρονα. Τι γίνεται με το εισόδημά του, πόσο εξαρτάται από τη γεωργία. Αν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την γεωργία, τότε, τότε δεν ξέρω κατά πόσο αυτό ο συλλογισμό που μα είπατε ισχύει 100%. Τι να σα πω, δεν είμαι ε, επαίων, επαίουσα στα γεωργικά, οικονομικά. Τόσο δεν ξέρω αν σα κατάλαβα καλά έτσι κι αλλιώ. Πρόεδρο. Απαντήστε μας, μια που έχουμε ακόμα λίγο χρόνο μέχρι χρόνο άλλη. Όχι, λέει η Μητρία, δεν είπα ότι θα πρέπει να, να, αναστείλουμε την κατάργηση. Ακόμη και στι αντισώμενε χώρες, μην πούμε υπάρχει και εκεί μια ομάδα καθαρά εξαγωγών και καθαρά εισαγωγών. Άρα είναι θέμα ισορροπίας. μέσω μακροπρόθεσμα θα πάνε καλά τα πράγματα για τις χώρες εκείνες και για τους Ευρωπαίου καταναλωτέ. Άρα, γι' αυτό σας λέω. Τι να σα πω, δεν ξέρω πόσο περισσότερο να το ξεκαθαρίσω. Θέλετε το λόγο, όχι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάτι να προσθέσει όχι προς το παρόν. Μάλιστα. Τότε για το ερώτημα το οποίο υποθέσατε και για το πώς θα συνεχίσουμε σε αυτές τις μελέτες βρισκόμαστε στη φάση των επαφών και θα αποφασίσουμε και θα σας ενημερώσουμε. Τώρα, βρισκόμαστε την αναμονή των άλλων εμπειρογνωμόνων Νομίζω ότι έρχονται τώρα οι ειδικοί για το επόμενο θέμα μας. Έρχονται από όλο τον κόσμο για αυτή τη τέταρτη ιστορική τράπεζα για την αποτελεσματικότητα των ε, ε, των ενισχύσεων θα γίνει αυτό στο Μπουσάν της Νοτιού Κορέας 29 Δεκάτου με 1η Δεκάτου του 2011 και πρόκειται να εξετάσουν την επιτευχθήσα πρόοδο παγκοσμίω όσον αφορά τον έχουμε περισσότερη αποτελεσματικότητα για την απτυξιακή βοήθεια και επίση πρόκειται να υπάρξουν δεσμεύσει, ούτω ώστε να μειωθεί η φτώχεια και να αναδειχθούν οι στόχοι της χιλιετίας για την ανάπτυξη. Εμείς είπαμε ότι θα κάνουμε μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας, άρα και σήμερα θα μπορέσουμε να βάλουμε τα θεμέλια για αυτή την έκθεση. Έχουμε την, τον, συνάδελφο Κριστιαν Ντανπρέντα που είναι ο εισηγητής και ήρθε να μας παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της έκθεσης του. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο που ήρθε και επίσης ε, και τον ειδικό ο οποίος θα έρθει όπου να είναι και θα βοηθήσει την συζήτησή μας, είναι ο κύριος Μπόντο Έλμερτς από την Eurodad. Donc nous accueillons Monsieur Elmer, qui est expert donc. Ah, ήρθε, ήρθε. Θα βοηθήσει τη συζήτησή μας, λέει πάλι ο Πρόεδρος. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο συζητείται τώρα μόνο σε επίπεδο επιτροπής. Και γι' αυτό δεν έχουμε καλέσει το Συμβούλιο, αλλά θα γίνει αυτό στην επόμενη συνάντηση τον Ιούλιο όταν παρουσιάσουμε την έκθεση. Je vais commencer par passer la parole à Christian Preda. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα πω δύο λόγια εν είδη προλόγου Πρώτα απ' όλα να σας υπενθυμίσω ότι η διεθνής κοινότητα θα συνεδριάσει στο Μπουσάνα από τις 29 Νοεμβρίου μέχρι την 1η ε, Δεκεμβρίου 2011 για να αξιολογήσει τις προόδους ε, στην εφαρμογή των δηλώσεων των Παρισίων του 2005 όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της βοήθειας καθώς επίσης ε, και την εφαρμογή του προγράμματο δράσης της άκρα του 2008. από τη στιγμή που πλησιάζουμε στην εκπνοή το 2015 θα αποφασιστεί από τους αρμοδίους το πλαίσιο των νέων μεταρρυθμίσεων όσον αφορά την ανάπτυξη. Η Επιτροπή, Ανάπτυξης αντιδρά για μία ακόμα φορά με έκθεση πρωτοβουλίας, όπως το υπενθυμίσατε άλλωστε, έτσι ώστε να καθορίσει τη βάση επί της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ζητήσει να εκφραστεί με μία φωνή η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το τέταρτο φόρουμ υψηλού επίπεδου. Πρέπει να πούμε ότι βάσει των πραγματικών στοιχείων διαπιστούται πρόοδος. Όμως η πρόοδος αυτής δεν είναι ικανή Εάν δεν γίνουν ε, πιο γρήγορες δράσεις ε, και πιο αποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις, δεν θα καταφέρουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας ε, που έχουμε, δηλαδή, τους στόχους που έχουμε στον τομέα αυτό, ούτε θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με το βήμα που θα θέλουμε θα πρέπει οπωσδήποτε να περάσουμε το απλό στάδιο της διαπίστωσης ε, και επομένως να προχωρήσουμε με απτές υλοποιήσεις έτσι ώστε να υλοποιηθεί πραγματικά η ατζέντα της αποτελεσματικότητας της βοήθειας. Σας προτείνω σήμερα να εστιάσουμε την προσοχή μας σε κάποιες σημαντικές προκλήσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιταχύνουμε την ε, διαδικασία της αποτελεσματικότητας της βοήθειας. Μεταξύ αυτών των στοιχείων νομίζω ότι πρέπει να αναφέρω πέντε που είναι τα σπουδαιότερα και που μπορούν να αποτελέσουν σημείο εκκίνησης στη σημερινή μας συζήτηση και βεβαίως ε, σημείο εκκίνησης όσον αφορά την ίδια την εκπόνηση της έκθεσης. Πρώτος, ε, πρώτη πρόκληση Πρώτη πρόκληση λοιπόν, ε, να διατηρηθεί ε, η οικονομική βοήθεια. Δηλαδή αυτό το τέταρτο φόρουμ θα πρέπει να θυμίσει στις ε, χώρες δωρητές την δέσμευσή τους να δίδουν το 0,7 του ΑΕΠ σε βοήθεια αναπτυξιακή και επίσης ε, να, ε, ότι πρέπει να σέβονται ε, τις αρχές του προγράμματος δράσης της ΔΑΚΡΑ. Δεύτερο, η αρχή της, οι αρχές της δημοκρατίας θα πρέπει να ε, ε, είναι μια προϋπόθεση εκ των ουκάνεφε για αυτή την αναπτυξιακή βοήθεια. Θα πρέπει να δοθεί επομένως μεγάλη σημασία ε, στην δράση της κοινωνίας των πολιτών, των, μέσος, των μέσων ενημέρωσης, του ιδιωτικού τομέα, αλλά και της διακυβέρνησης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο στη νέα αρχιτεκτονική της βοήθεια, το σημείο αυτό είναι καινούριο, αλλά βεβαίως θα πρέπει να δοθεί και η απαραίτητη αρρωγή έτσι ώστε να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές ε, να βελτιώσουν την νομοθετική τους δομή. Euh, Τρίτη μεγάλη πρόκληση. Ε, καταμερισμός της εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρέτησε το 2006 την, τον κώδικα ε, συμπεριφοράς ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τον καταμορισμό εργασίας και διαπιστώσαμε ότι δεν είχαν εφαρμοστεί και δεν εφαρμόζονται ακόμα οι αρχές αυτές. Δεν δίνεται μέσω της εφαρμογής των αρχών αυτών η μονάχα η δυνατότητα να εξοικονομηθούν πάρα πολλά χρήματα μέχρι 6 δις, αλλά ε, μπορεί να δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση κινητήριος ρόλος εις ε, την προετοιμασία του τέταρτου φόρουμ και την επιτυχή του έκβαση. Τέταρτη πρόκληση οι σχέσεις ε, με τους νέους χορηγούς, η ανάβηση νέων χορηγών, των οποίων η προσέγγιση δεν διέπεται ακόμα από τις ευρωπαϊκές αρχές δίνει την δυνατότητα για ένα νέο χώρο συνεννόησης έτσι ώστε να υπάρξει διαφάνεια ε, και ε, προώθηση στις σχέσεις αυτές γιατί διαφορετικά κινδυνεύουμε να έχουμε ένα σύστημα βοήθειας δύο ταχυτήτων από τη μία πλευρά την ε, παραδοσιακή μορφή που προσπαθεί από τη ρητορική, από τα λόγια να περάσει στις πράξεις και ε, η άλλη προσέγγιση όπου ο καθένας θα προχωράει με το δικό του τρόπο, με το δικό του βήμα, τις δικές του διαδικασίες και τις δικές του πολιτικές. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντική η τέταρτη πρόκληση. Πέμπτη πρόκληση και τελευταία θα πρέπει να έχουμε προσέγγιση στοχευμένη στα αποτελέσματα. Ε, βάση δηλαδή των ε, ε, αποτελεσμάτων και βάση της αιρεσιμότητας θα πρέπει να προχωρήσουμε. Ο ρόλος Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά αυτή την έννοια είναι πάρα πολύ σημαντικός γιατί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη βάσει τη συμφωνία της ΑΚΡΑ ε, ε, έχει ε, δώσει στους χορηγούς να καταλάβουν ότι εκ των αποτελεσμάτων θα κρίνεται η βοήθεια. Γενικώ μπορούμε να πούμε ότι ε, οπωσδήποτε θα πρέπει οποιαδήποτε προσπάθεια για την καλύτερη αποτελεσματικότητα της βοήθειας να περνάει μέσα από συνολικές πολιτικές. Γιατί το πλαίσιο του ΩΣΑ δεν μπορεί να εξαντλήσει ε, το θέμα της ανάπτυξης και επομένως θα πρέπει όλοι οι πρωταγωνιστές να συντονίσουν τις δράσεις τους έτσι ώστε να γίνει πραγματικά αποτελεσματική η βοήθεια. θα πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε πολιτικές απαντήσεις και συνολικές απαντήσεις γιατί διαφορετικά κινδυνεύουμε να επαναλάβουμε τις αποτυχίες του παρελθόντος. Αυτά ήθελα να πω κυρία Πρόεδρε εν είδη προημίου για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα της αποτελεσματικότητας της βοήθειας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρέντα, λέει Πρόεδρος. Οπωσδήποτε μας δώσατε έτσι μια ιδέα του τι ε, θα ε, ακολουθήσει. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Έμερς από την Eurodad. Okay, thank you very much for giving me the opportunity to speak here today. Ε, ε, λέγομαι Έλμες από την Eurodat και μιλώ εξ ονόματος της Concord που είναι η συνομοσπονδία των Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των Αναπτυξιακών Μη Κρατικών Οργανώσεων. Έχουμε συνεργαστεί με άλλες οργανώσεις από τον Νότο, με διεθνή συνδικάτα και με άλλες οργανώσεις και έχουμε αναπτύξει, τις θέσεις μας <clears throat> σε συνεργασία με <clears throat> τις άλλες αυτές οργανώσεις ε, από τον Νότο και ούτω καθεξής. Προ δύο εβδομάδων λάβαμε από τον ΟΟΣΑ την έκθεση αξιολόγησης της δήλωσης των Παρισίων. Τα πιο σημαντικά συμπεράσματα είναι ότι χρειάζεται περισσότερη αλλαγή, αλλά ότι χρειάζεται και περισσότερος χρόνος, αλλά και περισσότερη πολιτική βούληση για την υλοποίησή τους. Αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν, άρα χρειάζεται παρακολούθηση της ατζέντα. Ήδη αυτά έχουν οδηγήσει σε βελτίωση της ποιότητας της βοήθειας, καλύτερη συνεργασία μεταξύ δωρητριών και απολυτριών χωρών. Έχουν αυξηθεί οι όγκοι της βοήθειας, διότι γνωρίζουμε όλοι ότι χρειάζεται να βελτιωθεί και η αποτελεσματικότητα της βοήθειας, ώστε να παραμείνει, να, να ε, συνεχιστεί η κίνηση αυτή. Το πιο σημαντικό, ωστόσο, κατά τη γνώμη μας, συμπέρασμα ήταν ότι η δήλωση των Παρισίων ζητούσε λιγότερα από τους δωρητές από ό,τι από τους απολύπτες, αλλά ταυτόχρονα οι δωρητές έκαναν και ειδικότερες προσπάθειες. Αυτά, σε αυτά οδηγεί ο συσχετισμός δυνάμεων Για παράδειγμα, η υποχρέωση να χρησιμοποιούν τα συστήματα των χωρών υποδοχής, που είναι υποχρεωμένες να ενισχύσουν τα συστήματά τους, ενώ οι δωρητές είναι υποχρεωμένοι να τα χρησιμοποιήσουν. Εδώ οι δωρητές απίτησαν πρώτα να βελτιώσουν τα συστήματά τους οι ε, χώρε, χώρες, αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι εν τέλει θα χρησιμοποιηθούν τα συστήματα αυτά από τους δωρητές. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι τώρα οι δωρητές οφείλουν να κινηθούν, σύμφωνα με την δήλωση των Παρισιών. Οι προσδοκίες μας τώρα από το επόμενο πρόγραμμα όπως βλέπετε και στη διαφάνεια χρειαζόμαστε ανάληψη περισσότερων δεσμεύσεων στα πλαίσια του Busan Compact και χρειαζόμαστε επίσης λογοδοσία ή και μάλιστα και μηχανισμούς επιβολής. Ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχθηκε ε, σε σχέση με την δήλωση του ΩΣΑ ότι πρέπει να περιληφθούν οι μηχανισμοί επιβολής, διότι από ό,τι φαίνεται υπάρχουν δεσμεύσεις αλλά δεν ε, υλοποιούνται. Είναι σημαντικό στην προσπάθεια να συμμετάσχουν νέοι δωρητές, καθώς επίσης και ο ιδιωτικό τομέας, αλλά αυτά ίσως οδηγήσουν σε αποδυνάμωση των δεσμεύσεων. Και βέβαια χρειάζεται και ε, ανάμειξη ε, πολιτικού, πολιτικά υψηλού επίπεδου για τις ε, μη κρατικέ οργανώσεις είναι σωστό να υπάρξει η λεγόμενη ownership από πλευρά των χωρών μελών. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στη λεγόμενη δημοκρατική συμμετοχή, η δημοκρατική κυριότητα, democratic ownership, στον διάλογο για την ανάπτυξη των πολιτικών με συμμετοχή των κοινοβουλίων και της κοινωνίας των πολιτών. Είδαμε και την δήλωση της Βουδαπέστης, της ε, Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, που ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή των βουλευτών και, της, και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για, τα, για τους σχεδιασμούς. Εδώ εντάσσεται και η η αρχή ότι δεν μπορεί να υπάρχει ε, κυριότητα της διαδικασίας από πλευράς των, ε, χωρών, των, ε, των χωρών εάν υπάρχουν, υπάρχει χαιρεσιμότητα η οποία επιβάλλεται έξωθεν πολλοί δωρητέ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβάλλουν όρου, αιρεσιμότητα δηλαδή, ότι δηλαδή ε, πρέπει να έχει διασφαλιστεί για παράδειγμα η μακροοικονομική σταθερότητα ε, στην βάση της ερεσιμότητας ε, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Επίσης να χρησιμοποιούνται τα συστήματα της απολύτρια χώρας ως πρώτη επιλογή. Οι πολίτες και τα κοινοβούλια των απολυτριών χωρών δεν μπορούν να ελέγξουν τις τη βοήθεια παρά μόνο η βοήθεια που έρχεται και ρέει μέσω των δικών του συστημάτων και εφόσον υπάρχει η δημοκρατική κυριότητα. Εν τέλει, η τεχνική βοήθεια που αυτό απαιτείται μονάχα για την αποτελεσματικότητα της τεχνικής βοήθειας, που τώρα είναι πολύ ευαίσθητο θέμα, διότι οι σύμβουλοι τώρα βρίσκονται στα κέντρα εξουσίας των αναψώμενων χωρών, δηλαδή σε Υπουργεία Ανάπτυξης κλπ. Αλλά ποιοι τους, ε, ποιοι τους προσλαμβάνουν αυτούς, ποιοι τους πληρώνουν αυτούς και το καθεξής, αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν είναι ακόμα ξεκαθαρισμένα. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι να δοθεί προτεραιότητα σε ντόπιε δημόσιες προμήθειες ώστε να, να δημιουργηθεί απασχόληση και δυνατότητα εργασίας δηλαδή επί τόπου. Δύο τρίτα των συμβάσεων ανατίθεται ακόμα σε επιχειρήσεις που έρχονται από το εξωτερικό. Και αυτό δεν έχει φτάσει στα βέλτιστα επίπεδα για την ώρα. Επίσης χρειάζεται και προβλεψιμότητα των ροών βοήθειας. Τα βλέπουμε, βλέπουμε ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει κάνει μια καλή αφιτερία αλλά η διαθεσιμότητα της βοήθειας μπορεί να εξεταστεί και από μια μακροοικονομική ε, πτυχή, σκοπιά μάλλον. Ο, μπαίνει ως νέος παράγοντας και ο ιδιωτικός τομέας. Υπάρχουν ε, δημόσιες ροές αλλά και ιδιωτικές ροές από χώρα προς νότον και θα ήταν σωστό το Μπούζαν να φροντίσει ώστε να τονωθεί ο ιδιωτικός τομέας. να γίνει όμως με πιο υπεύθυνο τρόπο και καλύτερα προσαρμοσμένος στις ανάγκες. Η διαφάνεια είναι σημαντική. Υπάρχει σχετική πρωτοβουλία που ωστόσο δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από όλους τους Ευρωπαίους δωρητές. Εδώ μπορεί επίσης να εξυπηρετήσει το Μπουσάν. Εν τέλει, έχουμε στην ε, διακήρυξη των Παρισίων και την πτυχή της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, αλλά δεν λέει, έχουμε ακόμα ξεκαθαρίσει για ποια αποτελέσματα μιλούμε. Μιλούμε για την υλοποίηση ανθρώπινων δικαιωμάτων, μιλούμε για την ισότητα μεταχείριση των φύλων, για την ε, αηφορία του περιβάλλοντος και όλα αυτά πρέπει να μπουν μέσα σε όλους τους τομείς από την επιλογή των δημοσίων προμηθειών μέχρι το monitoring. Ο κέριος ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξακολουθεί να παίζει ε, τον σημαντικότερο ρόλο ε, στην βοήθεια, αν και ίσως έχει χάσει κάπως ελκυστικότητα τα τελευταία χρόνια, αλλά νομίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει το παράδειγμα, να ηγηθεί δια του παραδείγματος, να ασκήσει πίεση σε άλλους να ακολουθήσουν, να έχει δηλαδή φιλόδοξη προσέγγιση. Ούτε μπορούμε να παίξουμε το παιχνίδι «Α, εγώ δεν εφαρμόζω τα προβλεπόμενα επειδή εσύ δεν τα εφαρμόζεις» και ούτω καθεξής αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει τα απαραίτητα, τα στο ευρωπαϊκό επίπεδο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ε, βοήθειας που βασίζεται σε ορισμένα απορίσματα του ε, Συμβουλίου Υπουργών Ανάπτυξης, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι το λειτουργικό ή το επιχειρησιακό πλαίσιο πρέπει να υπάρχεται σε ένα μηχανισμό παρακολούθησης. πολύ σημαντικό ακόμη είναι η πολιτική δέσμευση στο Μπουζάν, τουλάχιστον σε υπουργικό επίπεδο. Και θα παρακαλέσω όλους και όλους να πιέσετε προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτά σας ευχαριστώ. Merci beaucoup pour cette... Ευχαριστώ πολύ για την εξαίρετη εισήγησή σας. Πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα να καλωσορίσω τους ε, τους καλεσμένους της συναδέλφου Κατρίν Γκρέζ από την περιοχή Μιντή Πυρενέ. Καλώς ήρθατε λοιπόν και ευχαριστούμε κυρία Γκρέζ που μας ε, φέρατε επισκέπτες. Είναι πάντα μεγάλη μας τιμή. Θα δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία Γκρέζ. Euh, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ που δεχτήκατε την ομάδα των επισκεπτών. Εγώ θέλω να πω δύο λόγια σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν από τους δύο προλαλήσαντες. Πρώτα απ' όλα για να τους ευχαριστήσω και για να πω ότι βεβαίως συμμερίζομαι απόλυτα την ιδέα ότι το Μπουζάν ε, θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή ε, για να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα της βοήθειας ε, και να αποτελέσει το έναυσμα για το νέο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων. Βεβαίω λέμε ότι θα πρέπει να εξορθολογιστεί το σύστημα, θα πρέπει να μιλάει η Ευρωπαϊκή Ένωση με μία φωνή και αυτό με βρίσκει απολύτως σύμφωνη. Αν τα καταφέρουμε αυτά, οπωσδήποτε θα είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια πάντα ε, θα είναι καλύτερη η κατάσταση από ότι οι ε, εθνικές αναπτυξιακές ε, πολιτικές ε, που γίνονται σε διμερές επίπεδο. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να επανέλθουμε σε αυτή τη βασική αρχή της αναπτυξιακής βοήθειας και δηλαδή να προσπαθήσουμε να αντιστρέψουμε μια λογική η οποία δεν είναι κατά την άποψή μου η καλύτερη. Πιστεύω ότι η ουσιαστικότερη ιδέα, τουλάχιστον έτσι βλέπει η ομάδα μου τα πράγματα, είναι το θέμα της κυριαρχίας. Εσείς εσείς αγαπητέ συνάδελφε μιλήσατε για την ε, λογοδοσία, για τον εκδημοκρατισμό, ε, δηλαδή μιλάμε περίπου για το ίδιο πράγμα. Η κοινωνία των πολιτών, ε, οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των χωρών αυτών θα πρέπει να χειρίζονται την αναπτυξιακή πολιτική. Νομίζω ότι αυτό είναι ε, ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο στην αντιμετώπιση μας και οδηγούμε έτσι στο επόμενο σημαντικό σημείο, ε, την ε, ερεσιμότητα. Ε, δηλαδή η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ε, επιβάλλουν εκ των έσω την ερεσιμότητα ε, και δεν δίνουν τη δυνατότητα στις χώρες να αποφασίσουν την οικονομική τους πολιτική οδηγούμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που ενδεχομένως είναι λίγο ταμπού. Παρόλα αυτά, εγώ τολμώ να πω ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτή η υποκρισία της ε, βοήθειας ε, που ε, περνάει και μέσα από τις δημόσιες προμήθειες. Ξέρουμε ε, πολύ καλά ότι σε αυτές τις χώρες, ε, τις ε, αναπτυσσόμενες, τελικά εμείς προωθούμε τις δικές μας εταιρείες. Εδώ θα επανέλθω σε κάτι που έχουμε ήδη από την αρχή της εντολής μας συζητήσει και εκπονήσει με την συνάδελφό μου κυρία Κέλλερ. Δηλαδή, σε τι χρησιμεύει να έχουμε ε, βοήθεια αναπτυξιακή και πολιτική τέτοιας αναπτυξιακής βοήθειας εάν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε εμπορική, γεωργική και αλλιευτική πολιτική που πηγαίνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Τολμάω να το πω. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε εγκάρσιες ε, πολιτικές και να έχουμε και εγκάρσιες συναλλαγέ απόψεων με τις άλλες επιτροπές. Αυτό ήθελα να πω. Και να σας πω τελειώνοντας ότι το Μπουζάν κατά την άποψή μου θα έχει καλά αποτελέσματα μονάχα εάν καταφέρουμε να μελετήσουμε σε βάθος αυτά τα σημεία τα οποία ανέφερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Γκρέζ. Η κυρία Θεοχάρους έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ να συγχαρώ τους δύο ομιλητές για την πολύ επικοδομητική, πολύ επικοδομητικές ομιλίες που έχουν κάνει και να εκφράσω την ελπίδα τη δική μου ότι στο Πουζάν θα γίνει αξιολόγηση της κοινή αναπτυξιακής πολιτικής και θα κινηθούμε προς ένα πιο αποτελεσματικό άξονα. Σύμφωνο με τους πέντε άξονες που έχει θέσει ο συνάδελφος μας στην ε, μελέτη που έχει κάνει. Ωστόσο θα έλεγα ότι είναι ξεκάθαρο πως είτε η βοήθεια που δίνουμε δεν έχει πραγματικά εκείνο τον όγκο που λέγεται ότι έχει, δεν είναι σε τέτοια ποσότητα για να φτάνει εκεί που πρέπει, είτε δεν είναι η κατάλληλη βοήθεια, είτε δεν γίνεται καλή χρήση της αναπτυξιακής βοήθειας από αυτούς που την δέχονται. Όποιο και είναι, όποια και να είναι η αιτία της αναποτελεσματικότητάς μας όλα αυτά τα χρόνια, σημαντικό είναι να αναθεωρήσουμε την πολιτική μας και να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό με εκπαίδευση, με γνώση, με μεταφορά δεξιοτήτων, γνωρίζοντας ότι η εκπαίδευση βοηθάει και την δημοκρατία και έτσι δεν θα έχει κανένα νόημα αυτό που λέγεται ότι η επιβολή πολιτικών από αυτόν που δίνει τη βοήθεια ε, πρέπει να είναι μια καθημερινή πρακτική. Γιατί η επιβολή πολιτικών συνδυάζεται πάντοτε με μείωση της κυριαρχίας αυτού που δέχεται την βοήθεια. Και δεν νομίζω ότι είναι κανείς που θα το ήθελε αυτό. Ε, βεβαίως την ίδια στιγμή που εμείς συζητάμε μεταξύ μας αν η βοήθεια που δίνουμε είναι ε, ανθρωπιστική ή αναπτυξιακή ή ε, αν πρέπει να δίνουμε βοήθεια και πώς, πρέπει να ξέρουμε ότι όλοι αυτοί που δέχονται τη βοήθεια δεν νοιάζονται καν τι είδους βοήθεια τους προσφέρουμε. Σας ευχαριστώ. Merci beaucoup. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κέλλερ. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω με όλα αυτά το είπε η Κατρίν και έχω να σας αναφέρω άλλα δύο θέματα. Δεν ξέρω, νομίζω τώρα κάποιοι που θέλουν να επικρίνουν, να εξετάσουν, να, αναλύσουν το τι κάνουν οι αναπτυσσόμενες κυβερνήσεις του ΣΥΠΗΝ, ε, χρησιμοποιούν πάρα πολύ το επιχείρημα της αποτελεσματικότητας ή αναποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής βοήθειας. Τελευταία, έχουν υποθεί πάρα πολλά για την αισθήση της ενίσχυσης, value for money, πιάσουν τόπο τα λεφτά κλπ. Όμως ε, Κοιτάξτε, στην πολιτική την αναπτυξιακή δεν βλέπει κανεί αποτελέσματα από το βράδυ στο πρωί, ούτε κάνουμε μέσα στην ίδια εκλογική θητεία. Είναι επομένω λίγο επικίνδυνο το να προσέχει κανεί να κρίνει το αποτελέσματο και, και, συνέχεια να, να επιμένει στο value for money, γιατί αυτό οδηγεί σε κοντόφθαλμη πολιτική, ενώ χρειάζεται μακρόπνοη ε, προοπτική. γιατί χτίζουμε και χτίζουμε σχολεία για το εξετάζουμε αυτό το μετράμε, όμως δεν μετράμε ακριβώς ποια είναι η επίπτωση στην παιδεία. Αυτό να το προσέξουμε πολλά κρατημέλια και, και, και η δική μου ίδια χώρα και η Κομισιόν να το προσέξει να μην ενδίδει στις σχετικές πιέσεις. Να την κάνουμε αποτελεσματική την ε, πολιτική και την ενίσχυσή μας αλλά μην κολλάμε. Τώρα όσον αφορά αυτούς τους αδειόμενους δωρητάς. Ε, Τα είπατε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο αυτό. Έχουμε αυτούς τους δωρητές. Είναι θέμα της αξιοπιστίας τους. Και γενικά το πόσο αξιόπιστη είναι αυτού του η αρρωγή. Αλλά το θέμα κατά πόσο εμείς μπορούμε να τους εμπλέξουμε. στι στις κινήσεις μας, στις πολιτικές μας, ε, άκρα και αυτά, και στον Μπουσάν ε, θα, θα παιχτεί πολύ το πόσο θα καταφέρουμε αυτούς τους δωρητές να τους εμπλέξουμε. Βέβαια είναι δύσκολο το θέμα, δεν έχουν ε, τόσο πολύ εμπλακεί ήδη. Άρα, τι να κάνουμε, τι κάνουμε και με τι συνέπειες. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό το να εμπλακούν και μάλιστα με τρόπο φιλόδοξο να μας εξηγήσει και η Κομισιόν βέβαια. Τι θέλει, τι επιδιώκει, τι θεωρείται ότι κατά τρόπο αποτέλεσμα που θα προκύψει από όλα αυτέ τι προσπάθειε που γίνονται και όσον αφορά του δωρητέ. Eh ε bien voilà, ça tombe bien. Je passe la parole à la Commission. Monsieur Grimaud. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Grimaud. Ε, ευχαριστούμε. Θεωρούμε ότι ήρθε την κατάλληλη στιγμή ε, αυτή η συνάντηση, μια που όπου να είναι, θα γίνει συνάντηση στο Μπουσάν και εμείς αποκρισταλώνουμε τις θέσεις μας και έχουμε το εξήχρονο διαγράμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν προβλέπει αρχές Σεπτεμβρίου την έκδοση ανακοίνωσης όπου θα διατυπώνει τις θέσεις της Ένωσης, στη συνέχεια δε, Οκτώβριο-Νοέμβριο θα το συζητήσει το Συμβούλιο. Άρα, η σημερινή συνάντηση ήρθε την κατάλληλη ώρα και έτσι θα μας βοηθήσει όλους να δημορφώσουμε απόψεις για το Μπουσάν. Επίσης, να δούμε τι έγινε και τι θα γίνει. Παρίσι, Άκρα και τώρα το Μπουσάν είναι θέματα που είναι στην διεθνή ατζέντα. Τώρα έχουμε τρεις άξονες στην διεθνή πολιτική της ανάπτυξης. Πρώτα πρώτα, στόχοι της χιλιτίας. Δεύτερο στοιχείο, χρηματοδότηση ανάπτυξης. Μοντερέι, Ντόχα και πάμε για την διάσκεψη του 2013 και τρίτο άξονα της σχέσης πολιτικής είναι αυτό που πέρασε από Παρίσι, άκρα και Παρίσι. Μιλούμε για αποτελεσματικότητα, δεν θα τα συζητήσουμε όλα. Στο Μπουσάν θα συζητήσουμε ε, τα θέματα της ε, διεθνούς διάταξης. Όλα αυτά τα θέματα συνδέονται το ένα με το άλλο, αλλά βασικά στο Μπουσάν θα συζητηθεί αυτό, η αποτελεσματικότητα της αντιξιακής βοήθειας. Εδώ και 10 χρόνια ξεκινήσαμε ε, αυτή την προσπάθεια και τώρα έρθει η ώρα του απολογισμού στο Παρίσι, συζητήθηκε στην Άκρα, στις γενικές γραμμές, υπήρξαν δεσμεύσεις και έχουμε συγκεκριμένους ε, δείκτες μετρήσιμους για να δούμε τι έγινε το 2010, πετύχαμε τους ε, στόχους μας και πόσο. Και έχουμε εδώ κάποιες υποχρεώσεις όσον αφορά τους εταίρους, τους δωρητές. Δεν νομίζω ότι έχουμε εδώ Έχουμε διαμόρφωση, συνένεση μεταξύ των μεν και των δε. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Αντίθετα με άλλες ε, συναντήσεις διεθνείς, όπου είχαμε αντιπαραθέσεις προχωρήσαμε συνετικά. Ορίσαμε υποχρεώσεις, αρχές, πράγματα που δεσμεύουν όλες τις πλευρές. Ο προλογισμός δείχνει ότι έχουμε σημειώσει πρόοδο, αλλά έχουμε και κάποιους στόχους που δεν πετύχαμε. Και επομένως, είπαμε ότι Προχωρούμε επί τη βάση των όσων διαπιστώσαμε και για τον Μπουσάν. Πρώτα-πρώτα έχουμε το θέμα του τι κάναμε στον την αποτελεσματικότητα, σε ποιο βαθμό τηρήσαμε τις προτεραιότητες. Είχαμε από Άκρα και Παρίσι 100 και πλέον δεσμεύσεις. Να δούμε τι καταφέραμε. Να, το πρώτο θέμα για τον Μπουσάν και κατόπιν να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στα πιο σημαντικά, να δούμε τι αποτελέσματα είχαμε και τι προτεραιότητες έχουμε. Η δημοκρατική επιτυχία του θέματος, όπως ο κ. Πρέντα, είναι πολύ σημαντικό. Το τι κάνουν τα κοινοβούλια. Η διαφάνεια επίσης, πάρα πολύ σημαντικό. Τον έφερε ο άλλο προσκεκλημένος. Να συνεχίσουμε αυτό το οποίο ξεκίνησε. Το είπε ο κ. Σέλμερς. τι έγινε με την ενίσχυση, τι δεδομένα έχουμε, τι αποτελέσματα πετύχαμε. Αυτό για το λένε και πιο σημαντικό και έχει να κάνει και με την δύσκολη οικονομική συγκυρία και επομένως κάθε ευρώ που ξοδεύεται στην ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να δικαιολογείται. Επομένως έχουμε εδώ πέρα ένα κίνδυνο και μια ευκαιρία. Όταν μιλούμε για αποτελέσματα δεν μιλούμε μόνο για βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα. Λέμε και για τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε πετύχει στις χώρες τους εταίρους μας. Τα αποτελέσματα που μαζί πετύχαμε με τους εταίρους μας. Σε Παρίσι και Άκρα συζητήθηκαν αυτά και είπαμε ότι θα αντίζουμε το σπαθιάς μας για να πετύχουμε και άλλα αποτελέσματα Δεύτερο μεγάλο θέμα ζήτησης στο Μπουσάν είναι η διεύρυνση της ατζέντα του και αυτό μας παραπέμπει στο θέμα των αναδειωμένων δωρητών και κατά πόσο αυτοί θα εμπλακούν άρα πρέπει να συμμετάσχουν όπως και η Κίνα έτοιμη, ενώ δεν ήταν μέχρι χτες. Άλλο θέμα, η υλοποίηση της αρχής της αποτελεσματικής βοήθειας και σε σχέση με την αλλαγή του κλίματος. Έχουν δει σχετικές δεσμεύσεις της Ένωσης, αυτό είναι μια πρόκληση για όλους. Και άρα να μην επαναλάβουμε τα σφάλματα του παρελθόντος. Νομίζω είμαστε αποτελεσματικοί όσον αφορά τη βοήθεια και σε αυτή την πολιτική. Άλλο όσον αφορά τα θέματα που πρέπει να προσθέσουμε στην ατζέντα είναι οι ευάλωτες χώρες. Και εδώ έχει να κάνει το θέμα αυτό με την αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης. συγχρηματοδότηση από ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στις χώρες εταίρους και έτσι να μπορεί η κοινωνία, οι εταίροι να συμμετάσχουν, να αναλάβουν τις ευθύνες τους όλοι σε αυτή την εργασιακή προσπάθεια. Τώρα όσον αφορά την ε, διακυβέρνηση, το πώς κάθε φορά θα υλοποιείται η σε πολιτική. Θα συζητήθηκαν και αυτά σε Παρίσι και Άκρα και είπαμε ότι θα πρέπει σε κεντρικό επίπεδο να γίνεται το ίδιο. Στον ΩΣΑ, στη αυτό, στις σχετικές ομάδες. Άρα τώρα θα πηγαίνουμε και πάλι τις μας στο πώς θα υλοποιείται η πολιτική όχι κεντροκατευθυνόμενα, αλλά επιτόπου στις εμπλεκόμενες χώρες. Στον Μπουσάν θα ζητηθεί αυτό και ίσως θα πρέπει να περικόψουμε την κεντροκατευθυνόμενη γραφειοκρατία και να βλέπουμε τις κάθε μιας χώρας τις ανάγκες. Και στο πιδάλιο κάθε φορά να είναι η εμπλεκόμενη χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Προτείνω τώρα να πάρει το λόγο εκπρόσωπος, ε, ένας από τους δύο εκπροσώπους της Eurodat, όποιος θέλει, για να απαντήσει. Comme Όποιος από τους δύο επιθυμεί. Okay, my name is Mayra Morococo. Mayra της ε, Action Aid International. παρακολουθούμε την διαδικασία αυτή από την πλευρά της κοινωνίας των πολιτών. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα σχόλια που κάνατε. Να πω όμως δύο σχόλια. Πρώτον, αναφέρεστε στην κατάργηση της οικονομικής αιρεσιμότητας. Υπάρχει όμως και ένα άλλο ερώτημα και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε σαφείς και όσον αφορά το σημείο αυτό. Ε, σε σχέση δηλαδή με τη νέα δεοντολογία της ε, βοήθειας θα πρέπει να αναφέρουμε και άλλους όρους ερεσιμότητας, ε, δηλαδή σε σχέση με τη διαφορά και τα ανθρώπινα, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Νομίζω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουμε υπόψη μας ε, και αυτήν την ερεσιμότητα και οπωσδήποτε θα πρέπει να δούμε κυρίως χώρες οι οποίες έχουν υπογράψει ήδη και επικυρώσει διεθνείς συμφωνίες ε, και σε αυτές τις χώρες οπωσδήποτε η κοινωνία των πολιτών ε, θα πρέπει να ελέγχουν κατά πόσον ε, η διακυβέρνησή τους εφαρμόζει αυτές τις συμφωνίες. Τώρα, η πολιτική διάσταση της ανάπτυξης, ε, δεν θυμάμαι την ακριβή διατύπωση, αλλά ε, οπωσδήποτε η συνθήκη της ε, Λισαβόνας ε, αναφέρεται συγκεκριμένα στα θέματα αυτά. πρέπει να αποφασίσουμε με ποιο τρόπο ε, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, γιατί έχουν ήδη αληφθεί υποχρεώσεις ε, και για αναπτυξιακούς στόχους. Επίσης, ε, το τελευταίο που θα σχολιάσω αφορά στο ζήτημα της ισότητας των φυλών και των φύλων συγγνώμη, και το τράφικινγκ. Όπως είπε και ο συνάδελφος, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε αποτελέσματα, αναπτυξικά, αναπτυξιακά αποτελέσματα. Και ε, βεβαίως δεν πρέπει απλώς να μετράμε πόσα σχολεία χτίζουμε, αλλά ε, να βλέπουμε τι επίπτωση έχουμε, τι αντίκτυπο έχουμε στην πραγματική κοινωνία και πόσο γίνονται σεβαστά τα οικονομικά αλλά και κοινωνικά δικαιώματα όλων των μελών της κοινωνίας. Ευχαριστώ. Μπορώ να πω και εγώ δύο λόγια, ναι. Η κυρία Γκρέτς μίλησε για ε, ε, συνεκτική πολιτική και συνοχή έτσι, όλων των πολιτικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε επίσης σε άλλα παρόμοια σημεία. Ναι, ε, συμφωνώ με όλα αυτά που ανέφεραν οι βουλευτές και οι Κομισιόν, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το Φόρουμ ε, Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχουν φόρα για την κλιματική αλλαγή. Δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα στο Φόρουμ για την ε, αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Επίσης υπάρχουν χώρες όπως η Κίνα, ας πούμε, ε, που δεν δέχονται πλήρως τα όσα είχαν αποφασιστεί και από τον ΩΣΑ για τα θέματα αυτά to speak about issues in the framework of the UN, so I would call on Νομίζω ότι ε, θα πρέπει να ζητήσω και εγώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει πιο σοβαρά υπόψη της τα όσα γίνονται στο αναπτυξιακό φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών. Κύριε Πρεντά, θέλετε το λόγο για να ολοκληρώσετε. Δεν σας βλέπω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εδώ είμαι, εδώ είμαι, δεν φεύγω. Πού να πάω. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους και μη για τις ε, παρατηρήσεις τους. Δύο λόγια ήθελα να κάνω σχετικά με τα σημεία τα οποία έφυξαν ε, οι κυρίες εκ δεξιών μου, που δεν είναι της δεξιάς, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Βρίσκονται στα δεξιά μου. Η ιδέα της κυρίας Γκρέζ, η ιδέα ε, αυτής της, ε, ε, της δημοκρατικής ας πούμε δικαιοδοσίας, λογοδοσίας, συγγνώμη. Βεβαίως, βεβαίως μας ενδιαφέρει αυτό. Είναι κάτι με το οποίο συμφωνούμε απολύτως. Η πολιτική ευθύνη βεβαίως βρίσκεται στην πλευρά, κατά την άποψή μου, των κυβερνώντων και επομένως θα πρέπει να καταναλώνεται με προσοχή γιατί διαφορετικά ε, εάν όλα περάσουν από την κοινωνία των πολιτών ε, ίσως ε, στρεβλωθεί και λίγο αυτή η ιδέα της αναπτυξιακής βοήθειας. Δεύτερον, μερικές φορές είναι γεγονός ότι είναι λίγο δύσκολο να, πει κανείς να κάνει κανείς συγκεκριμένες μετρήσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα. Και όσον αφορά και όσον αφορά αυτήν την ε, λογική των αποτελεσμάτων όσον αφορά αυτή την ιδέα των αποτελεσμάτων δηλαδή, ε, θα πρέπει να είμαστε και λίγο υπομονετικοί. Πάντως, συμφωνώ κυρία Κέλλερ μαζί σας, ε, δηλαδή συμμερίζομαι και εγώ την ανησυχία για την Κίνα. Είναι γεγονός ότι η θέση της ε, Κίνας πηγαίνει πλέον προς την πλευρά των αναδειωμένων ε, δωρητών. Θα δούμε, όπως είπε και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, ε, πώς θα εξελιχθεί η Κίνα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να περιμένουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα περιμένω με πολύ μεγάλη ε, προσμονή την έκθεση και το φόρουμ και την έκθεση που θα λάβει χώρα στην επόμενη... τον, τον επόμενο μήνα. Τώρα θα κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση, μάλλον την γνωμοδότηση του συναδέλφου Νόρμπερτ Νόιζερ, ε, όσον αφορά το στάδιο εφαρμογή στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση για την Κεντρική Ασία. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μα, τον κύριο Νόιζερ, για να μα παρουσιάσει αυτήν την γνωμοδότηση. Κύριε Νόιζερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε, κυρία Πρόεδρε. Όντως αυτή η γνωμοδότηση για την Κεντρική Ασία είναι μια γνωμοδότηση η οποία ε, αφορά ε, έκθεση για την οποία ε, επί της ουσίας είναι υπεύθυνη η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εμείς θα ασχοληθούμε μονάχα με το θέμα της ανάπτυξης θα πω δύο λόγια για τις χώρες της Κεντρικής Ασίας πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα η κατάσταση των χωρών αυτών είναι ακόμα πάρα πολύ περίπλοκη και όσον αφορά το κοινωνικό και το πολιτικό ε, επίπεδο. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις συνήθως είναι δικτατορικές, απολυταρχικές ε, και είναι κατάλοιπα το, ε, ε, του σοβιετικού οικοδομήματος και δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για την οικονομική ευημερία των πολιτών τους, τουλάχιστον όχι τόσο όσο ενδιαφέρονται για να κρατήσουν την θέση τους. Το είδαμε άλλωστε αυτό σαφώς και στην ακρόαση από τις απόψεις που εξέφρασαν διάφοροι ε, πολιτικολόγοι και ειδική σε θέματα Κεντρικής Ασίας. Θα ήθελα να επανέλθω τώρα σε δύο ε, σημεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για την γνωμοδότηση την οποία εκπονούμε. Ε, πρώτον, ο πόλεμος στο Αφγανιστάν και δεύτερον, η ενεργειακή αυτάρκεια, μάλλον προμήθεια ε, της Ευρώπης όσον αφορά το Αφγανιστάν το 2014 θα αποσυρθούν από ό,τι φαίνεται ε, τα στρατεύματα ε, και επομένως ε, οι χώρες της Κεντρικής Ασίας φυσικά θα έχουν πολύ ωφεληθεί από την κρίση αυτή. Γιατί οι υποδομές μεταφορών αλλά και οι προμήθειες του ΝΑΤΟ ε, έδωσαν την δυνατότητα στις χώρες αυτές να εμπλακούν στις διαδικασίες αυτές. Ε, βασιστήκαμε λοιπόν στις χώρες αυτές ε, για να συνεχίσουμε την παρουσία μας στο Αφγανιστάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι έκλεισε τα μάτια ε, όσον αφορά ε, και τα όσα συνέβησαν στο Ουσμπεκιστάν το 2005. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, δεν ε, αν έκανε λίγο τα στραβά μάτια, δεν επέβαλε κυρώσεις. Επίσης υπάρχει το ζήτημα ε, του South και του Ναμπούκο ε, και το θέμα λοιπόν της ε, ενεργειακής προμήθειας της Ευρώπης. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί καμιά φορά όταν μπερδεύονται τα οικονομικά με τα πολιτικά και όταν στη μέση υπάρχει και η πολιτική για το Αφγανιστάν τα πράγματα μπερδεύονται πολύ. Zunächst mal, dass wir gegenüber den θα πρέπει να Έχουμε πλέον τελείως διαφορετική, διαφοροποιημένη προσέγγιση απέναντι στις χώρες ε, της ε, Κεντρικής Ασίας. Θα πρέπει να πούμε και στην Κομισιόν ότι τα προγράμματα βοήθειας θα πρέπει να είναι ξέχωρα τα μένα από τα δε. Υπάρχει η αναπτυξιακή βοήθεια για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, για τον έλεγχο των συνόρων, ε, και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία βεβαίως δεν αμφισβητούνται ε, ουδόλως γιατί θα βοηθήσουν και θα ανακουφίσουν την κοινωνία των πολιτών. Και οπωσδήποτε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει τον ρόλο της κοινωνίας των ε, πολιτών. Θα πρέπει να ενδυναμωθεί η θέση των τοπικών ε, κοινωνιών καθώς επίσης ε, και ε, των τοπικών αρχών γιατί στο δομημένο διάλογο αυτές παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η ανεπτυξιακή μας πολιτική θα πρέπει να λάβει υπόψη της όλα τα στοιχεία αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Κίνιτσεν η οποία είναι εισηγήτρια για την ΑΦΕΤ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο για την έκθεσή του με την οποία συμφωνώ Και εγώ ασχολούμαι με την έκθεση αυτή που αφορά τι χώρε τη Κεντρική Ασία και όντω, ε, όπω τα είπε, υπάρχει εδώ μεγάλο έλλειμμα όσον αφορά τη κυβέρνηση, ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία κλπ. Παρ' όλα αυτά, συμφωνώ και με εσά που είπατε ότι χρειάζεται μια διαφοροποιημένη προσέγγιση. Μια που υπάρχουν διαφορετικέ ανάγκε σε κάθε χώρα από αυτέ. Όλε αυτέ που εμεί τι λέμε συνολικά Κεντρική Ασία, α πούμε στο Κυργιστάν, Κυργισία, έχουμε την πρόεδρο τη χώρα ε, η οποία κατά κάποιο τρόπο αποτελεί μια χτίδα ελπίδα μέσα στην όλη αυτή η περιοχή. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε επίση και μια διάκριση όσον αφορά την χορήγηση τη ε, ενίσχυση. Τα ξέρουμε όλα αυτά, όπω τα είπατε στην έκθεση, όσον αφορά το Αφγανιστάν. Για πιο συγκεκριμένα, όχι, συγγνώμη, το Ουσβεκιστάν, λέει ο όσον αφορά το, το, του στόχου για το 2005 που είπαμε, για τα γεγονότα που έγιναν τότε. Ε, αυτά που είναι το 2005 είναι πάρα, πάρα πολύ σοβαρά και εμεί όταν πάμε εκεί θα συζητήσουμε πάνω σε αυτά και είπαμε ότι δεν καθόμαστε στο τραπέζι να τα συζητήσουμε εάν δεν γυρίσουν σελίδα. Δεν ήμασταν πάρα πολύ αποτελεσματικοί σε σχέση με τα όσα είχαμε πει, γιατί δεν ε, ίσχυσαν οι κυρώσει Τα ξέρει ο κ. Νόιζερ και γι' αυτό είναι υπεύθυνη η Γερμανία, η οποία ακριβώ προβληματίζεται για το τι γίνεται με τα γερμανικά στατεύματα τα οποία βρίσκονται στο Αφγανιστάν, στα σύνορα. Ε, το Ουσμπεκιστάν, ε, τότε που υπήρχε αυτή η προστριβή, όλα αυτά. Κατά τα συμφωνώ με τον κ. Νόιζερ, επίση από την κοινωνία των πολιτών για το Καζακστάν. Εκεί ήρθαμε σε επαφή με κάποιου φορεί που ε, μα είπαν ότι δεν είναι φυσιολογικό το να μην έρχεται σε επαφή μαζί μα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπαμε και εδώ υπάρχει ένα κενό και αυτό θα πρέπει να το ψάξουμε, α πούμε, σε, όπου είναι δυνατόν να έχουμε την κοινωνία των πολιτών. Όπου γίνεται στο Καζακστάν, στην Τουρκμενία, α πούμε, δεν γίνεται. Στην Κυριακή επίση γίνεται και άρα θα πρέπει οπωσδήποτε να αφουγκραστούμε την των πολιτών και γι' αυτό συμφωνώ με τα όσα είπατε σχετικά. Ε, Επίση, όσον αφορά την κατανομή τη βοήθεια, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ανέφερε για σήμερα το πρωί στην Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διότι είπαμε ότι έχουμε κάποιες μη κυβερνητικέ οργανώσεις που ξεσκεύασε ένα σκάνδαλο ε, γιατί έχουμε αυτά τα 3 εκατομμύρια ευρώ για αυτό το ίδρυμα που όμως απευθεία ε, ε, διοικείται και χειρίζεται η κόρη του Προέδρου στο Ζουμπεκιστάν, 3,7 ε, εκατομμύρια και όλα αυτά τα χειραγωγεί αυτή η κυρία τα ελέγχει άμεσα. Ε, οπότε είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει πραγματικά επαγρύπνηση όσον αφορά την χορήγηση κατανομή της βοήθειας σε αυτήν την χώρα. Όλα αυτά ελπίζω να μπουν στην έκθεση. Ευχαριστούμε λοιπόν και τώρα για το λόγο ο κύριος Γκοράνσα. Ευχαριστώ, συνάδελφε Νόιτζερ. Πάρα πολύ αξιολογική έκθεση. Δεν έχω να πω κάτι συγκεκριμένο σαν παρατήρηση. Εκτός από κάποια σημεία τα οποία νομίζω δεν θα πρέπει να ζητηθούν και για την έκθεση αυτή, αλλά και για τις τυχόν επόμενες εκθέσεις. Χρειάζεται μια στρατηγική, διαφοροποιημένη προσέγγιση. Και αυτό θα είναι η απάντηση στην περιπλοκότητα της κατάστασης που αντιμετωπίζουμε. Σε τεχνικό, τεχνοκρατικό επίπεδο θα πρέπει να το προσέξουμε τι γίνεται με την ενεργειακή πολιτική, ακόμα και για το Ιράν, σαν αφορά την προμήθεια της ενέργειας. Παντού θα πρέπει να προσπαθούμε να έχουμε μια πολιτική διαλόγου. Έστω και σε τεχνικό επίπεδο. Και αυτό είναι καλύτερο από το τίποτα. Τώρα μια παρατήρηση για τις δυσκολίες της εμπλοκής και των πολιτών. Το είπε και η τι γίνεται όσον αφορά τον προπολισμό της Ένωσης και τους πόρους αυτούς που πήγαν στο Ίδρυμα που ελέγχει η κόρη του Προέδρου. Να μην είμαστε υποκριτές. Δεν μπορούμε να κάνουμε την πολιτική μας χωρίς κίνδυνο. Αν κανείς θέλει μηδενικό κίνδυνο, τότε θα πρέπει να αδρανήσει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα με τις ε, τοπικές ε, αρχές, ούτε με την κοινωνία. Άρα, θα πρέπει να είμαστε θωρακισμένοι όσον αφορά τις ε, επικρίσεις. Να παίρνουμε το ρίσκο, να εξηγούμε στον κόσμο τι γίνεται. Γιατί ε, άμα απλά ε, γκρινιάζουμε, άμα απλά αποθούμε τις δυσκολίες, ε τότε δεν θα κάνουμε τίποτα με αυτές τις χώρες που υπάρχει χαοτική κατάσταση, υπάρχει πρόβλημα διακυβέρνηση. Να βοηθήσουμε την Κομισιόν να ασχοληθεί με το πρόβλημα. Να μας τα πει η Κομισιόν, να μας ζητήσει τι γίνεται, μέχρι ποιο είναι. Μπορούμε να δείξουμε αυτή την εμπιστοσύνη, κοινωνία των πολιτών, μη κυβερνικές οργανώσεις, να δώσουμε την σκητάλη σε εκείνες. Σου δώσουμε την εντολή Οπότε είναι το θέμα πάρα πολύ λεπτό, δύσκολο. Θα πρέπει να δούμε το ότι πιο εύκολο είναι το αποδεκτές με οργανώσεις από τα θεσμικά όργανα. Αυτά. Επομένως, Πάρα πολύ καλά τα είπε ο κ. Νόιζερ και θα το στηρίξουμε. Θα δώσω το λόγο στην ε, Επιτροπή, κ. Ζαγκλούλ Κουεντά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή κ. Νόιζερ και την εισηγήτρια της ε, Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Πρέπει να σας πω ότι η Κομισιόν δέχεται ε, τα στοιχεία τα οποία προτείνει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ε, ο εισηγητής ε, της Επιτροπής Ανάπτυξης όσον αφορά τις χώρες της Κεντρικής Ασίας. Νομίζω ότι σωστό είναι να βασίσουμε ε, την ε, προσπάθειά μας και την βοήθειά μας ε, στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλα τα άλλα στοιχεία τα οποία ανέφερε και ο εισηγητής. Άλλωστε η πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει από το 2007 εκεί βασίζεται. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι ε, συμφωνούμε με την διαφοροποιημένη προσέγγιση ε, προς τις ε, πέντε χώρες της περιοχής ανάλογα με το δυναμικό τους και την ήδη αναπτυξιακή τους πορεία. Ξέρετε ότι υπάρχουν χώρες όπως το Κυργιστάν, ας πούμε, που έχουν πολύ πιο δομημένα προγράμματα, ενώ το Ουσμπενιστάν το Ουσβεκιστάν και το Τουρκμενιστάν είναι λίγο αντίθετη περίπτωση και το Καζακστάν επίσης διαφορετική γιατί το, το οικονομικό δυναμικό είναι τελείως διαφορετικό και δεν απαιτεί τόσο μεγάλη αναπτυξιακή βοήθεια. Μεγάλη διαφοροποίηση λοιπόν. Θα ήθελα παρόλα αυτά να σκεφτείτε ότι η διαφοροποίηση αυτή δεν θα πρέπει να ανασχέσει την προσπάθειά μας ε, να στηρίξουμε περιφερειακές ε, πολιτικές ε, που ενθαρρύνουν τις χώρες της περιοχής να συνεργαστούν ε, σε θέματα ας πούμε, διαχείρισης ε, συνόρων ή κοινή διαχείρισης υδάτινων πόρων. Επομένως, πέρα από τις διαφοροποιήσεις που πρέπει να έχουμε απέναντι στις πέντε αυτές χώρες, θα πρέπει να στηρίξουμε ε, ενοποιημένες περιφερειακές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες. Τρίτον, η διαφοροποίηση, η διάκριση μεταξύ των ε, μηχανισμών. Ε, ε, από τη μία πλευρά λοιπόν ο μηχανισμός σταθερότητας και από την άλλη το DCI. Βεβαίως όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και ε, συμπληρωματικότητα των στόχων. Ας πούμε, όσον αφορά το κράτος δικαίου, κάποιες ε, δράσεις έχουν ξεκινήσει με το εργαλείο σταθερότητος, όμως μπορούν ε, να συνεχιστούν με τα θεματικά του, του άλλου σκέλους και του άλλου μηχανισμού και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε πιο αποτελεσματικά και πιο βιώσιμα προγράμματα στις ε, χώρες αυτές, έτσι ώστε να τις βοηθήσουμε να, να βοηθήσουν, να, να βελτιώσουν τη λειτουργία του δικαϊκού συστήματος, του δικαστικού συστήματος, νόμου καθώς επίσης και του Κοινοβουλίου. Συμπληρωματικότητα λοιπόν των εργαλείων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί ε, το αποτέλεσμα. Βεβαίω θα πρέπει να ενισχυθεί και η κοινωνία των πολιτών. Όπως έλεγε όμω και ο κύριος Γουμέντ, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να συνεργαστεί κανείς με την κοινωνία των πολιτών σε χώρε, ε, οι οποίε δεν είναι ελεύθερες και επομένως η κοινωνία των πολιτών δεν έχει πάντα τη δυνατότητα ελεύθερα να εκδηλωθεί. Βεβαίω εμεί έχουμε προγράμματα τα οποία στηρίζουν την ανάδυση της ε, κοινωνίας των πολιτών. Ε, και στο Κυργιστάν και στο Ουσβεκιστάν έχουμε τέτοια προγράμματα. Επίσης, συνεργασία και ε, συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Ε, βεβαίως θέλουμε να έχουμε καλύτερη σύνδεση και με τις περιφερειακές και τοπικές δομές. Αυτά ήθελα να πω κυρία Πρόεδρε όσον αφορά τα στοιχεία τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. σα ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο ξανά στον κύριο Νόιζερ, εάν θέλει να κάνει τις τελικές τους, τα τελικά του συμπεράσματα. Σα ευχαριστώ για τι παρατηρήσει σα. Νομίζω ότι περίπου συμπλέουμε. Ορισμένα πράγματα ίσως τα βλέπουμε κάπως διαφορετικά. Όπως είπα, η δική μας Επιτροπή είναι αρμόδια μόνο για την αναπτυξιακή συνεργασία και δεν θα πρέπει να υπερβούμε τα όρια αυτά. Θα είμαι ευγνώμων για εισδήποτε προτάσεις. Αυτά, αρχούμε σε αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Υπενθυμίζω ότι την 23η Ιουνίου στις 5 το απόγευμα λήγει η προθεσμία υποβολής τροπολογιών και ότι η ψηφοφορία θα λάβει χώρα την 24 η Σεπτεμβρίου. Υπό τα διάφορα έχουμε κάτι? Όχι. Επομένως, επόμενη συνεδρία τη Επιτροπής Ανάπτυξης θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες ε, στις 12 Ιουλίου από τις 9.30 μέχρι τις 12.30 και από τις 3 μέχρι τις 6.30 καθώς επίσης και την 13η Ιουλίου από τις 9 μέχρι τις 12.30. Σας υπενθυμίζω πάντως ότι ε, έχει κληθεί η Επιτροπή μας να συμμετάσχει σε ένα σεμινάριο σήμερα το απόγευμα που έχει ε, συνδιοργανωθεί με την Επιτροπή Περιβάλλοντος με θέμα την ευρωπαϊκή απάντηση στις καταστροφές και εγώ εκλήθην να συντονίσω το πρώτο τμήμα του σεμιναρίου. Σας περιμένουμε λοιπόν πολυπληθείς, θέλουμε να είναι πολυπληθής η παρουσία σας, 2,5 PH1002 PHS ένα α λοιπόν 002. Σας ευχαριστώ πολύ και για μία ακόμα φορά λυπούμε γιατί δεν έχουμε μεγάλη παρουσία των βουλευτών σε αυτές τις συνεδριάσεις. Ευχαριστώ πολύ.